Hello to everybody. I think it's... Καλημέρα σε όλους. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Hello to everybody. Καλημέρα σε όλους. Έχουμε πολλά Σήμερα το πρωί έχουμε την συνεδρίαση της Επιτροπής και θα ακολουθήσει η συνεδρίαση συντονιστών. Με πολύ σημαντικούς προσκεκλημένους σήμερα δύο υπουργού της ε, Φιλανδίας ε, λόγω της Φιλανδικής Προεδρίας. Θα ήθελα να τους καλωσορίσω λοιπόν. Για να ξεκινήσουμε πρέπει να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Υπάρχουν προτάσεις ή ενστάσεις στην ημερήσια διάταξη που έχουμε προτείνει. Θα θεωρήσω ότι την έχουμε εγκρίνει. Έχω να κάνω μια ανακοίνωση που θα μας ε, χαροποιήσει όλους. Σήμερα μπορείτε να ακούσετε διερμηνία σε όλες τις γλώσσες. πρέπει να εγκρίνουμε τη πρακτικά των συνεδριάσεων της 10ης, 15ης και 18ης Ιουλίου. Νομίζω ότι έχετε λάβει όλοι μέσω email τα πρακτικά και γνωρίζετε σε ποια έγγραφα αναφερόμαστε. Μπορούμε λοιπόν να τα εγκρίνουμε. Θεωρώ ότι έχουν εγκριθεί. Ευχαριστώ. Πάμε στο κύριο πρόγραμμα για τη σημερινή συνεδρίαση. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους ε, προσκεκλημένους μας. Τον Υπουργό Απασχόλησης της Φιλανδίας, κύριο Τίμο Χαράκα, και την κυρία Άινο Κάισα Πέκονεν, Φιλανδή Υπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας. Καλωσορίσατε στην Επιτροπή μας. Πριν δώσω το λόγο στους προσκεκλημένους μας, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι μεγάλο πλήθος μέλων της Επιτροπής μας εξέφρασε την επιθυμία να υποβάλει ερωτήσει στους προσκεκλημένους μας. Αυτό θα γίνει σε δύο γύρους. Ο πρώτος γύρος θα είναι ο γύρος των συντονιστών. Θα πάρω λοιπόν τα ονόματά τους για το ΕΛΚΑ Είναι ο κ. Ντένι Ράτκα. Για τους Σοσιαλιστέ, η κυρία Γκάμπι Μπίσοφ. Για το ΑΡΗ e, η κυρία Ντράγκο Πίσλαρου. Για τους πράσινου, κυρία κύρα Πέτρα Χάνσεν. Για το ID ο κύριος Φρανζαμέ. Για το ECR η κυρία Ασμπέτα Ραφάλσκα. Και για την ΚΟΕ ο κύριος Νικολάη Βίλεμψεν. Είστε όλοι εδώ. Ωραία. Όχι. Μάλιστα, ε, πράσινη. Ναι, καλημέρα. Η κυρία, κυρία Πίτερ Χάνσεν δεν είναι εδώ, αλλά εγώ είμαι συνσυντονίστρια Κατρίν Λαγκζίβεν, οπότε θα μπορούσα εγώ να την αντικαταστήσω. Ωραία, το δέχομαι, λέει πρόεδρος. Πάμε τώρα. Θα έχουμε λοιπόν αυτό τον πρώτο γύρο που θα δώσω το λόγο στους συντονιστές και θα ακολουθήσουν ε, οι απαντήσεις όλες μαζί σε όλες σας τις ερωτήσεις και μετά θα έχουμε το δεύτερο γύρο με έναν πραγματικά πολύ μεγάλο κατάλογο μελών της Επιτροπής. Θα ανακοινώσω και τις ώρες και το χρόνο μάλλον. Οι συντονιστές θα έχετε ο καθένας δύο λεπτά. Σας παρακαλώ να τηρήσετε το χρόνο γιατί θέλω να πάρουν το λόγο όλα τα μέλη της Επιτροπής που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετέχουν στη συζήτηση. Θα είμαι λοιπόν πολύ αυστηρή με τους χρόνους. Ξεκινάμε λοιπόν δίνοντα το λόγο στους φιλάνδου προσκεκλημένους και πρώτος ο κύριο Χαράκα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να σας συγχαρώ κύριε Πρόεδρε και να συγχαρώ και τους αντιπροέδρους για την εκλογή τους. Ελπίζω ότι η συνεργασία μας θα είναι επικοδομητική για το καλό της Ευρώπης. Πρέπει να πω ότι για μένα προσωπικά αυτή η στιγμή είναι πολύ σημαντική. Το να βρίσκομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πριν από 25 χρόνια είχα την ευκαιρία να εργαστώ εδώ ε, πριν η Φιλανδία γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή πριν από ένα τέταρτο του αιώνα. Ε. Οπότε είναι μεγάλη μου χαρά σήμερα το ότι βρίσκομαι εδώ ως υπουργό για να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα της φιλανδική Προεδρίας, της τρίτη φιλανδική Προεδρίας. Φυσικά τα πράγματα δεν είναι όπως ε, στις δύο προηγούμενες ε, προεδρίες το 1999 και το 2006. Όπως γνωρίζετε βρισκόμαστε σε μια μεταβατική εποχή θεσμικά Συνεχίζουμε τις εργασίες ε, της Ρωμανικής Προεδρίας όσον αφορά το νομοθετικό κομμάτι, αλλά έχουμε την ευκαιρία και θα έλεγα μάλιστα και την υποχρέωση να έχουμε μια επικοδομητική συνεργασία ε, και ένα στρατικό πρόγραμμα με την επόμενη Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Και αυτό για το μέλλον της Ευρώπης. Θα πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι, ε, να δείξουμε βούληση. Αυτό θέλουν από εμάς ε, οι Ευρωπαίοι πολίτες. Όπως γνωρίζετε, οι στόχοι της Φιλανδικής ε, Προεδρίας θα μπορούσαν να συνοψιστούν με τα έξι λόγια. Μια βιώσιμη Ευρώπη, ένα βιώσιμο μέλλον. Θέλουμε να διασφαλίσουμε μετάβαση προς μια ουδέτερη κλιματικά οικονομία και βιώσιμη από κοινωνική άποψη. Θα επιμείνουμε στις θεμελιώδεις αξίες ε, το σεβασμό του κράτους δικαίου, την ανταγωνιστικότητα, μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς. Θέλουμε επίσης να ενισχύσουμε τη θέση της Ευρώπης ε, στην παγκόσμια σκηνή και να είμαστε πρωτοπόροι σε κλιματικά θέματα. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα προκύψει ε, μια στρατηγική βιώσιμης ε, ανάπτυξης και χωρίς αποκλεισμούς. Θέλουμε επίσης να εφαρμόσουμε το στρατηγικό πρόγραμμα που υιοθέτησε τον Ιούνιο το Συμβούλιο. Θέλουμε να επιμείνουμε επίση στο πρόγραμμά μα στην κοινωνική ισότητα, στο πλαίσιο αυτό τη μετάβαση ε, σε μια πιο κλιματική οικονομία. Όσον αφορά την απασχόληση, ε, στην ΕΠΣΚΟ πριν ε, λίγους, ε, λίγες εβδομάδες συζητήσαμε για έναν καθαρό πλανήτη. Αυτή τη μετάβαση, δηλαδή προς μια ουδέτερη οικονομία όσον αφορά τα κλιματικά θέματα. Οι υπουργοί θεωρούν ότι είναι σημαντικό η μετάβαση αυτή να γίνει τάχιστα, χωρίς αποκλεισμούς ε, κοινωνικούς και με δίκαιο τρόπο. Πρέπει να επικαιροποιούμε διαρκώς τις γνώσεις μας και να επιμένουμε στον κοινωνικό διάλογο ούτως ώστε να διασφαλιστεί αυτή η ισότιμη μετάβαση. Στον επιχειρηματικό κόσμο θα πρέπει να στραφούμε ψηφιακό, στην ψηφιακή τεχνολογία χωρίς να ξεχνάμε την κατανομή της εργασίας και την κοινωνική βιωσιμότητα. Οι εργαζόμενοι πρέπει διαρκώς να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ένα καλό επίπεδο απασχόλησης. Αυτά τα θέματα προβλήθηκαν στη διάσκεψη που διοργανώσαμε στο Ελσίνκι τον Ιούλιο. Επικεντρωθήκαμε στην ψηφιοποίηση, στην διαβίου μάθηση και στην εκ νέου αναδιοργάνωση της εργασίας. Και θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις αυτές στο πλαίσιο του ΕΠΣΚΟ. Επιπλέον θέλουμε να διασφαλίσουμε ίσες δυνατότητες για όλους. Αυτό είναι ουσιώδου σημασίας, διότι η ισότητα είναι σημαντικό κομμάτι ε, της πολιτικής, της κοινωνίας και της οικονομίας. Σήμερα βλέπουμε τεράστιες αλλαγές στον κόσμο της εργασίας ε, που συνεπάγονται νέες προκλήσεις. Οι συνθήκες εργασίας, η ασφάλεια στην εργασία πρέπει να διασφαλίζονται ακόμη και υπό αυτές τις νέες ε, μορφές εργασίας. Δεν μπορούμε να αφήσουμε κανέναν στο περιθώριο. Κυρίες και κύριοι, όπως γνωρίζετε, από νομοθετική άποψη η Φιλανδική Προεδρία δεν θα έχει και πολλά να κάνει. Θα χρειαστεί να βασιστούμε στο άριστο έργο που έχει ήδη γίνει από την Αυστρία και από τη Ρουμανία κατά τη διάρκεια των δικών τους Προεδριών. Εμείς απλά θα διασφαλίσουμε τη συνέχεια αυτών των σημαντικών θεμάτων. Μετά έχουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus, για τα οποία θα πρέπει να διασφαλίσουμε μια κοινή θέση. Επίσης θα χρειαστεί να ρυθμίσουμε ζητημάτα δημοσιονομικά το Συμβούλιο έχει καταλήξει σε μια μερικώς κοινή θέση όσον αφορά το ESF ε, και το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Θέλουμε να συνεχίσουμε τις προσπάθειες στο πλαίσιο τριλόγων με το δικό σας κοινοβούλιο, με το κοινοβούλιο εδώ, ε, στο διάρκεια της προεδρίας μας. Οι επιχειρήσεις και οι μισθωτοί έχουν να αντιμετωπίσουν παγκόσμια ανταγωνιστικότητα. Από δικής μας πλευράς ε, έχουμε εκπονήσει τη διακήρυξη για την επέτειο του Παγκόσμια Οργάνωσης Εργασίας. Ε, θέλουμε να διασφαλίζονται σωστοί κανόνε εργασίας. Θέλουμε να διασφαλίζεται ε, η ποιότητα της εργασίας σε όλη ε, την αλυσίδα παραγωγής. Ε, όλα αυτά για την εκατοστή επέτειο του Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Η Φιλανδία μελετά αυτή τη στιγμή τα συμπεράσματα του Συμβουλίου όσον αφορά την ενίσχυση, την ενδυνάμωση της απασχόλησης. Θέλουμε να διασφαλίσουμε την κοινωνική ισότητα και να βελτιώσουμε επίσης και τις δεξιότητες των μισθωτών, των εργαζομένων. Επίσης πρέπει να επιμείνουμε στις ε, δυνατότητες εργασίας από ψυχολογική άποψη, από σωματική άποψη και να ενισχύσουμε τις γλωσσικές δυνατότητες και τις λοιπές δεξιότητες. Αυτό θα εξαρτηθεί φυσικά από την εκπαίδευση αλλά και από ε, τις ανάγκες των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Θέλουμε να συζητήσουμε περί της ανακοίνωσης της Επιτροπής που αφορά τι αποφάσεις που λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία στον τομέα τη κοινωνικής πολιτικής. Επίσης πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις συνθήκε εργασία ε, στις ε, τρίτε χώρες. Όλα αυτά μέσω προτάσεων της Κομισιόν που εμείς θα συζητήσουμε με τα διάφορα κράτη-μέλη. Επίση, θέλουμε να συζητήσουμε την υλοποίηση του πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων στο επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στα διάφορα κράτη-μέλη. Θα συζητήσουμε για τι διάφορε προκλήσει ε, στον τομέα τη κοινωνική πολιτική και τη πολιτική απασχόληση. Επίση, ε, επί του θέματο αυτού, θα διοργανώσουμε στι 9 Δεκεμβρίου ένα δείπνο για του υπουργού, όπου θα καλέσουμε επίσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους κοινωνικούς εταίρους καθώς και μέλη της δικής σας επιτροπής. Στο νομοθετικό μέτωπο τα κράτη-μέλη έχουν να υλοποιήσουν διάφορες οδηγίες. Εμείς από πλευρά μας θα πρέπει να ενισχύσουμε την υλοποίηση αυτών των διαφορών νομοθετημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις. Όσον αφορά την κινητικότητα των εργαζομένων, θα συνεχίσουμε τις εργασίες που ξεκίνησε η Μπρατισλάβα. Πιστεύω ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε μια ικανοποιητική κινητικότητα των εργαζομένων δίκαιη και βέβαιη. Λαμβάνοντα φυσικά πάντα υπόψη τα δικαιώματα των εργαζομένων. Θεωρούμε ότι ο κοινωνικό διάλογο είναι κάτι πολύ σημαντικό θα λαμβάνουμε συνεπώς υπόψη τις ε, ε, γνώμες των κοινωνικών εταίρων. Στις 16 Οκτωβρίου μάλιστα θα έχουμε μια τριμερή σύνοδο κορυφής. Ε, έχουμε την πρόθεση να προσκαλέσουμε σε αυτή τη σύνοδο και ευρωβουλευτές. Αυτά κυρία Πρόεδρε. Θα κλείσω εδώ και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις των βουλευτών. Παρακαλώ. Thank you very much, Mr. Minister, for your speech. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Τηρήσετε και το χρόνο σας. Η κυρία Πέκονεν τώρα. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλω κι εγώ να σας ευχαριστήσω για την οργάνωση της ακρόασης αυτής. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να είμαι εδώ και να μιλώ μαζί σας για την προεδρία της χώρας μου και την βελτίωση της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης που νομίζω ότι αποτελεί ξεκίνημα μιας πολύ χρήσιμης περίοδου συνεργασίας που θα συνεχιστεί και μετά την προεδρία μας. Η συνεργασία μας θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε μία ένωση δηλαδή όπου οι πολίτες θα λειτουργούν καλά και κυρίως καλύτερα από ό,τι πριν. Αυτή είναι η δουλειά μας ως, εκπρόσωποι, ως εκπροσώπων των πολιτών. Η... Από αυτό θα εξαρτηθεί και η επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά. Ο συνάδελφος μίλησε για τις προτεραιότητες της Προεδρίας από την οπτική των πολιτικών απασχόλησης και της αγοράς εργασίας. Εγώ θα σας μιλήσω για τις ε, πρωτοβουλίες το δικό μου κομμάτι, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ασφάλιση και υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Στην ε, πλατφόρμα του Πρωθυπουργού μας, εμφανίζεται σαφώς μία δήλωση. Η ευημερία των πολιτών είναι ο κύριος στόχος. Το μέλλον και η ευημερία των πολιτών μας είναι ο κρογωνιαίος λίθος του προγράμματός μας. Η οικολογική και κοινωνική βιωσιμότητα που αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες της χώρας. Σε αυτό περιλαμβάνεται το βασικό εισόδημα, η μόνιμη κατάρτιση, που αποτελούν θεμέλια για μια ισχυρή και δίκαιη δράση της κυβέρνησης. Η οικονομία είναι για το λαό, όχι το ανάποδο. Ο στόχος μας είναι να έχουμε πολίτες που είναι ευχαριστημένοι από τη δουλειά τους, που είναι ευτυχισμένοι με την επαγγελματική τους επιλογή και που έχουν αποκτήσει δεξιότητες που μπορούν να προσφέρουν τώρα στην κοινωνία. Αυτό είναι η βιωσιμότητα και η ευθύνη μας, να αναλάβουμε, να φροντίσουμε όλους. Όσους, ιδίως όσους δεν αισθάνονται δυνατοί, άτομα που γερνάνε, δεν πρέπει να αποκλείσουμε κανέναν νέο. Να μεριμνήσουμε ώστε οι οικογένειες υποστηρίζονται και μπορούν να μεγαλώσουν με δίκαιο και ισότιμο τρόπο τα παιδιά τους. Να φροντίσουμε ούτως ώστε αυτή η, η ανάπτυξη να μην γίνεται εις βάρος της φύσης και των πεπερασμένων πόρων της γης μας. Αυτές είναι οι αξίες που διέπουν την, την πολιτική μας στην κυβέρνηση αλλά και την προεδρία μας όπως σας είπα. Οι προτεραιότητες μας είναι οι κοινέ αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κράτος δικαίου, μια ένωση που είναι πιο ανταγωνιστική και πιο συνεκτική κοινωνικά, που είναι πρωτοπόρος στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, που ενδιαφέρεται για την ασφάλεια των πολιτών τας με έναν ολιστικό τρόπο. Αυτό είναι η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης και αυτό είναι η δική μου αρμοδιότητα. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό πέραν της κοινωνικής πολιτικής να ασχοληθούμε με τον όπου η Ένωση έχει ισχυρές εξουσίες και άρα όπου που αποτελούν προτεραιότητα για μας. Η Ευρώπη πρέπει να φανεί ότι προωθεί την ευημερία των πολιτών συνολικά. Μιλώ για τις οικονομικές πολιτικές, τις πολιτικές της εσωτερικής αγοράς, η, η προσέγγιση αυτή την καλούμε, την προσέγγιση αυτή την καλούμε συχνά η οικονομία της ευημερία. Και αυτό είναι αυτό που διέπει την Προεδρία μας. Ο στόχος είναι η προσέγγιση αυτή να είναι στο κέντρο των μελλοντικών στρατηγικών της ε, Ένωσης και να αποτελέσουν το επόμενο βήμα για την ανάπτυξη της κοινωνικής διάστασης Ευρώπης. Η ευημερία της οικονομίας στηρίζεται στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων και ο στόχος μας είναι η σωστή και πλήρης εφαρμογή του πυλών αυτού. Σύμφωνα με τις συνθήκες, ο κύριος στόχος, ένας κύριος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προώθηση της ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών. Συχνά η οικονομική ανάπτυξη ωστόσο παίρνει μεγαλύτερη προτεραιότητα, που σημαίνει ότι μερικές φορές ενδεχομένως ξεχνάμε ότι η ευημερία είναι ένας βασικός στόχος της Ένωσης ο στόχος ωστόσο της οικονομικής ανάπτυξης δεν είναι αποκλειστικός. Αντίθετα, είναι, οι δύο στόχοι είναι αμοιβαία ενισχυόμενοι. Οι πολιτικές ευημερίες βελτιώνουν την παραγωγικότητα, την κοινωνική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Φροντίζουμε όμως ταυτόχρονα να μην αποκλείεται κανένα σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα και εξασφαλίζουμε ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι είναι ασφαλής και ότι κάποιος φροντίζει για αυτούς. Η μία λειτουργική κοινωνική πολιτική αποτελεί το θεμέλιο μιας βιώσιμης ε, ανάπτυξης. Και βέβαια ο στόχος μας είναι να εφαρμόσουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης εν ώψη του 2030, όπως υιοθετήθηκαν από τον ΟΗΕ. Όχι όμως εις βάρος της ευημερίας των πολιτών. Μία οικονομία της ευημερίας επιτρέπει στους πολίτες να αισθάνονται καλά. Δεν χρειάζομαστε νέες αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο, ούτε καν νέες δομές. Απλώς χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τις υφιστάμενες δομές και τις υφιστάμενες αρμοδιότητες. Για παράδειγμα, μπορούμε να κάνουμε πιο αποτελεσματική την πρόσβαση της ε, Ένωσης, την εμπλοκή της Ένωσης σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής, στον χώρο εργασίας, ισότητας δικαιωμάτων. Ο στόχος μας είναι το Συμβούλιο, να έχουμε συμπεράσματα του Συμβουλίου τον Οκτώβριο για την ευημερία των πολιτών και να υιοθετήσουμε συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ε, ισότητα και την οικονομική ανάπτυξη καθώς και την προστασία και υγιεινή και ασφάλεια το Δεκέμβριο. Θα θέλαμε να κάνουμε και μια συζήτηση για τα θέματα αποκλεισμού στην Ευρώπη. Υπάρχει ακόμα πολύ μεγάλο, υπάρχουν ακόμα πάρα πολλέ διακρίσει αυτή τη στιγμή. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, όπω τόνισε και ο συνάδελφο κ. Χάρακα, Έχουμε πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη του Υπουργείου. Ένα βασικό ζήτημα είναι και τα, η προσέγγιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης μετά την πολύ καλή δουλειά που έκανε και η Ρουμανική Προεδρία. Πρόκειται για ένα σύνθετο εξαιρετικά τεχνικό φάκελο και θέλουμε να προχωρήσουμε όταν ακούσουμε και τη θέση του Κοινοβουλίου για το ζήτημα αυτό. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και περιμένω ανυπόμονα τις ερωτήσεις σας, τις οποίες θα προσπαθήσω να απαντήσω μαζί με τον κύριο Χαράκα, ανάλογα με τα χαρτοφυλάκια του καθενός μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που ε, τηρήσατε το χρονομιλία σας και σας ευχαριστώ και για τις πληροφορίες που μας δώσατε, κυρία Υπουργέ. Το λόγο έχουν οι συντονιστές στον πρώτο γύρο της συζήτησης. Ο κάθε ένας από τους 7 συντονιστές έχει δύο λεπτά για να θέσει την ερώτησή του. Ξεκινάμε λοιπόν από το ΕΛΚ και τον κύριο Ντένις Ράτκε. Κυρία Πρόεδρε, κυρία, κύριοι Υπουργοί, ε, συνάδελφοι, σας ευχαριστώ θερμά για την επισκόπηση της Προεδρίας σας που μας δώσατε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια από τα θέματα που αναφερθήκατε. Είπατε ότι θέλετε μία συνάντηση κορυφής των κοινωνικών εταίρων, ε, μία πρωτοβουλία που επικροτώ. Στη συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ συχνά, ε, ξεχνιέται ότι η κοινωνική οικονομία της αγοράς μπορεί να λειτουργήσει μόνο με τους ε, κοινωνικούς εταίρους. Και μάλιστα η πολιτική χρειάζεται πολύ λίγες διορθωτικές κινήσεις ε, να κάνει. Γι' αυτό επικροτώ την ε, πρωτοβουλία σας. Βέβαια η Προεδρία σας ε, έρχεται σε δύσκολους καιρούς. Ε, έχουμε την απειλή του σκληρού ε, Brexit που έχει αυξηθεί τώρα με την εκλογή του Μπόρις Τζόνσον. Εσείς πώς θα προετοιμαστείτε προορατικά για τις κοινωνικές επιπτώσεις που θα πλήξουν τους Ευρωπαίους πολίτες που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ίσως θα μπορούσατε να πείτε λίγα λόγια για το θέμα αυτό. Επίσης αναφέρθηκαν ε, τα ακόμη εκρεμή ζητήματα ε, της προηγούμενης ε, θητείας, η διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη, το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης και άλλα. Μήπως μπορείτε να μας πείτε τι σκέφτεστε. Επίσης, ο προϋπολογισμός είναι σημαντικό θέμα, η κοινωνική Ευρώπη χρειάζεται και χρήματα. Και Μία τελευταία παρατήρηση. Χθε ήμουνα στην ε, Ήτρε. Ε, εκεί το θέμα που δεσπόζει είναι η αλλαγή του κλίματος. Ε, δεν έχω αντίρρηση εδώ στην Επιτροπή μας να μιλάμε για τις κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Το θέμα όμως είναι πότε θα ξεφύγουμε από αυτές ε, τις αόριστες δηλώσεις ότι ναι, πρέπει να ξεφύγουμε από την κατάσταση, λαμβάνουμε υπόψη μας σοβαρά το θέμα. Πρέπει κάποια στιγμή να προχωρήσουμε σε ε, συγκεκριμένα μέτρα. Στην δική μου περιφέρεια αυξάνεται ο φόβος ε, σχετικά με τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος. Θα ήθελα παρακαλώ τις παρατηρήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπίσοφ. Σας ευχαριστώ πολύ που μοιραστήκατε τις ιδέες σας και τους στόχους της Προεδρίας σας μαζί μας. Προσβλέπουμε στην Προεδρία σας και χαιρόμαστε που έχετε θέσει την αηφορία σε όλες τις διαστάσεις, ε, κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά. Και νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον να εξετάσουμε τι είναι η αηφόρος, η κοινωνία με ισότητα. Πιστεύω ότι οι ανισότητες είναι ένα από τα θέματα κλειδιά αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα θέμα με το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε. Επίσης, ε, αηφόρος επιχείρηση. Τι ακριβώς είναι αυτό. Ε, πρέπει να έχουμε καλή υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Πρέπει να έχουμε καλή συμμετοχή των εργαζομένων και γι' αυτό επικροτώ το ότι εστιάζεται στον κοινωνικό διάλογο και θα ήθελα να ξέρω τι σκοπεύετε να κάνετε για να ενισχύσετε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις διότι όπως γνωρίζετε τα τελευταία χρόνια αποδυναμώθηκαν ε, και αυτή ήταν μία από τις προκλήσεις που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω τον κοινωνικό πυλώνα, τον πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. ο πατέρας του κοινωνικού πυλώνα αποχωρεί, έχουμε μια μεταβατική περίοδο, χρειαζόμαστε νέους γονείς για τον κοινωνικό πυλώνα και χρειαζόμαστε ε, συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για να τον εφαρμόσουν και να ενισχύσουμε την ε, εμπιστοσύνη των πολιτών. Να τους δείξουμε ότι αυτό δεν ήταν απλά μια κοινή υπόσχεση, ήταν ε, το θεματολόγιο για τα επόμενα χρόνια. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω ποια είναι τα σχέδια σας, ώστε ο πυλώνας αυτός να γίνει σχέδιο δράσης. Και επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στην ψηφιοποίηση που βρίσκεται στο κέντρο του προγράμματός σας. Ε, είναι τεράστια η πρόκληση και θα πρέπει να διαμορφώσουμε πολιτικά ε, την όλη διαδικασία. Σημαντικό θα είναι εδώ να έχουμε επικαιροποίηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των κοινωνικών δικαιωμάτων και να ε, περάσουμε σε μια νέα εποχή στον χώρο της εργασίας και θα ήθελα να Θα ήθελα να ξέρω και ποιες είναι οι προσδοκίες σας ε, και το λόγο τώρα έχει ο κύριος Πίσλαρου. Θα παρακαλούσα την κυρία Λάνιεν Ζήπεν να αρχίσει να ετοιμάζεται να πάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, στο όνομα της ομάδας Renew Europe θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις εισηγήσεις σας και για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Είναι μεγάλη μας χαρά να σας καλωσορίσουμε εδώ. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την επιθυμία μου για ισχυρή συνεργασία μαζί σας κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Η πολιτική μας ομάδα, όπως λέει και το όνομά της, θέλει να ανανεώσει την Ευρώπη. Πιστεύουμε στην μία ενωμένη Ευρώπη, ε, όχι μόνο ενωμένη ε, όσον αφορά το Βορρά, τον Νότο, την Ανατολή και τη Δύση, αλλά και μια ενωμένη κοινωνία. Πιστεύουμε ότι ο φαύλο κύκλος του κοινωνικού αποκλεισμού θα πρέπει να σπάσει και να έχουμε μια ε, ανταγωνιστική οικονομία που να κινείται με βάση μια συμμετοχική κοινωνία. Η οικονομία της ευημερίας ε, είναι κάτι με το οποίο έχει ασχοληθεί η ΩΣΑ έχει τον ε, δείκτη καλύτερης ε, ζωής, για παράδειγμα. Πιστεύουμε στην αγορά, πιστεύουμε όμως ε, και στην κοινωνική ένταξη. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή πάνω από 25 εκατομμύρια παιδιών στην Ευρώπη ζουν υπό συνθήκες φτώχειας ή ε, δεν ε, απολάβουν ε, επαρκών κοινωνικών παροχών. Η φιλανδική κοινωνία, όπως γνωρίζουμε, επικεντρώνεται στις ευκαιρίες σε μια εξειδικευμένη αγορά εργασίας. Πώς συνδυάζονται όλα αυτά με το υπόλοιπο πρόγραμμα της Προεδρίας σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εκ μέρους της ομάδας μας πώς θα χρησιμοποιήσετε την Προεδρία σας ε, για να προωθήσετε την εγγύηση για τα παιδιά, κάτι που υπογράμμισε και η Ursula von der Leyen. Πώς ε, θέλετε να προωθήσετε τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ποιες είναι οι συγκεκριμένες πολιτικές που θα προωθήσετε τη στιγμή που δεν έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες μας ε, για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη. Σας ευχαριστώ πολύ, προσλέπω στη συνεργασία μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ η κυρία Κάτριν Και παρακαλώ, ε, κυρία Φρανσεμέ να ετοιμάζεστε να θέσετε την ερώτησή σας. Η κυρία Λάγγεν-Ζήπεν, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, κυρία Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, ακούσαμε πολλές ε, καλές παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ θερμά για τις εισηγήσεις σας. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρεις τομείς αναφέρατε ότι κανένας δεν επιτρέπεται να μείνει πίσω. Όλοι θα πρέπει να συμμετέχουν, να έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στην εργασιακή ζωή, άσχετα από το πόσο καλά εξειδικευμένοι είναι. Θα πρέπει πάντα να έχουν ευκαιρίες μετεκπαίδευσης. Υπάρχουν όμως κάποιοι που παρόλα αυτά δεν τα καταφέρνουν στην ε, Γερμανία ε, αντιμετωπίζουν δυσκολίες άτομα με αναπηρίες που συχνά ζουν και εργάζονται σε προστατευμένα ιδρύματα και δεν έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν και να εργαστούν αυτόνομα. Αναφερθήκατε στις διακρίσεις στον χώρο εργασίας. Επίσης, η φτώχεια είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ο προλαλής σας μίλησε για την φτώχεια των παιδιών. Ε, έχουμε τους άστεγους. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό θα μπορούσε να πλήξει τον καθένα μας. Το να βρει κανείς στέγαση είναι πρόβλημα στην Ευρώπη, είναι δύσκολο. Η Φιλανδία ε, είναι πρωτοπόρος όσον αφορά το πρόγραμμα Housing First που έχει να κάνει με άστεγους ανθρώπους που πέφτουν θύματα διακρίσεων στην αγορά εργασίας, σε άστεγους, άνεργους. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω τι θα κάνετε για αυτούς τους ανθρώπους κατά τη διάρκεια της προεδρίας σας. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Φρανς Ζαμέ. Και παρακαλώ και η κυρία Ραφάλσκα να ετοιμαστεί για την ερώτησή της. Ναι, κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, άκουσα πολύ προσεκτικά τις ε, προτεραιότητες ε, της Φιλαδικής Προεδρίας της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγώ διαφωνώ. Δεν υπάρχει καμία επαφή με την πραγματικότητα όσον αφορά τις φιλοδοξίες σας και θέλω να αναφέρω δύο αρχές που λέτε εσείς μια βιώσιμη Ευρώπη, ένα βιώσιμο μέλλον, την κινητικότητα των Ευρωπαίων εργαζομένων και τα καλύτερα ταλέντα του τρίτου κόσμου που πρέπει να ενθαρρύνονται να έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με άλλα λόγια, κοινωνικό dumping, μαζική μετανάστευση, θα τα ενθαρρύνετε στη διάρκεια της Προεδρίας σας. Η κινητικότητα των Ευρωπαίων εργαζομένων σήμερα ονομάζεται απόσπαση εργαζομένων. Είναι ένα νέο όνομα και στη δική μου τη χώρα, τη Γαλλία, Ουσιαστικά μιλάμε για μια εκμετάλλευση των Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης για να μην μιλήσουμε για τον αθέμητο ανταγωνισμό. Αυτή η φημισμένη κινητικότητα έχει οδηγήσει ένα σωρό κόσμο σε χρεοκοπία ε, και ένα σωρό κόσμο στην ανεργία. Τα καλύτερα ταλέντα του τρίτου κόσμου ακούγεται πολύ όμορφο. Έρχονται στην Ευρώπη και ουσιαστικά ε, εκμεταλλεύονται τους δικούς μας πόρους, διατηρώντας τις δικές τους χώρες επανάπτυκτες. Και μάλιστα γιατί τέτοιε προτεραιότητες. Εδώ και δεκαετίες θέλετε η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει μια οικονομία γνώσης και κοινοτομία. Σε τι χρησιμεύουν λοιπόν όλες αυτές οι προθέσεις αν φέρνουμε από αλλού τα μυαλά τα οποία θα έπρεπε να μας δίνουν τα δικά μας ε, ε, πανεπιστήμια, η Μπολόνια, η Σορβόνη, η Οξφόρδη όλα αυτά δεν χρησιμεύουν σε τίποτα. Και με άλλου ε, ευρωπαϊκού λαού δεν μπορούμε παρά να καταγγείλουμε, να θλιβόμαστε για αυτέ του τοξικού στόχου μια τέτοια πολιτική και του επικίνδυνου στόχου, τον φιλελευθερισμό και τη μετανάστευση, την υποστήριξη τη μετανάστευση. Κάτι που μα απομακρύνει από την οικονομία τη ευημερία που εσεί λέτε ότι υποστηρίζετε. Κυρία Ραφάλσκα, έχετε εσεί το λόγο. Και κύριε Βίλεμσον, παρακαλώ προετοιμαστείτε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργή. Οι προτεραιότητες ε, της ε, Φιλανδικής Προεδρίας ε, μου φάνηκαν ενδιαφέρουσες. Είναι πολύ ευγενείς και πιστικές προτεραιότητες. Αϊφόρος Ευρώπη, αϊφόρο μέλλον, αϊφόρος ανάπτυξη, κοινωνική ισότητα όλα ωραία και καλά, αλλά η ε, ερώτηση είναι πότε θέλουμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Όσον αφορά το στόχο, μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε. Αλλά πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και μπρος. Παρά είναι γενική η συζήτησή μας. Μιλάμε για τον κοινωνικό διάλογο ε, και θέλουμε να τον προωθήσουμε ε, που ήδη έχουμε λήψεις στον τομέα αυτό. Θέλουμε να έχουμε ε, κοινωνικό θεματολόγιο, αλλά και αυτό έχει διαφορετική μορφή σε κάθε χώρα. Η κυρία Υπουργό μίλησε για τα κοινωνικά ζητήματα, μίλησε για τους στοχότερους, για τους αποκλεισμένους. Όσον αφορά την φτώχεια, φτώχεια των παιδιών, των γονιών, των αποκλεισμένων. Πώς ε, θα αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Η, η, ε, η μας γυράσκει. Αυτές είναι οι μεγάλες προκλήσεις. Η, η ε, μίλησε και για ε, κοινωνικές υπηρεσίες προς όλους. Γιατί υπηρεσίες μιλάμε. Ε, υπηρεσίες προς ηλικιωμένους, προς παιδιά και η οικονομία της ευημερία τι ακριβώς είναι. Μπορείτε να μας δώσετε πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Πιστεύω ότι στην παρούσα φάση θα έπρεπε ήδη να έχουμε προχωρήσει περισσότερο. Θα έπρεπε να συζητάμε συγκεκριμένες νομοθετικές ε, πράξεις. Υπάρχουν νέες τεχνολογίες στην αγορά εργασίας μας ε, που αποτελούν πρόκληση, διότι θέλουμε να διατηρήσουμε τις θέσεις απασχόλησής μας, ε, θέλουμε να προωθήσουμε τη μετεκπαίδευση και μεγάλο πρόβλημα είναι ε, και η κοινωνική ανισότητα. Σας ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Βίλουμσεν. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. ευχαριστούμε τους Φιλανδούς φίλους που βρίσκονται εδώ εκ μέρους της ομάδας της αριστεράς. Θα ήθελα να συγχαρώ την όμορφη χώρα σας, τη Φιλανδία, για την προοδευτική της ε, κυβέρνηση και εκ μέρους της ομάδας της αριστεράς ε, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που συμμετέχουν και οι φίλοι μας ε, από την Φιλανδική Αριστερά στη Συμμαχία. Σας έχω δύο ερωτήσεις. Πολλοί Ευρωπαίοι εργαζομένοι βλέπουν να υποβαθμίζονται οι συνθήκες εργασίας τους. Συνάδελφοι από άλλες χώρες της Ευρώπης πληρώνονται ανεπαρκώς, τους κακομεταχείριζονται, υποβαθμίζονται ε, με κοινωνικό τάμπινγκ ε, και οι συνθήκες και οι μισθοί. Και η ερώτησή μου είναι η Φιλανδική Προεδρία θέλουμε να εργαστεί υπέρ του κοινωνικού πρωτοκόλου όπως προτείνεται. Δεύτερον η Βαντερ Λάιεν έχει ανακοινώσει ότι θα υποβάλει μια πρόταση για έναν κατώτατο μισθό πανευρωπαϊκό. Αυτό φυσικά θα βοηθήσει ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον μπορεί κανείς να ζήσει με αυτά τα χρήματα αλλά στις ε, χώρες του Βορρά μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στο μοντέλο αγοράς-εργασίας με τις συλλογικέ συμβάσεις. Οπότε η ερώτησή μου είναι η Φιλανδική Προεδρία ε, θα διασφαλίσει ότι ο κατώτατος μισθός πανευρωπαϊκά δεν θα θέσει σε κίνδυνο το μοντέλο των βόρειων χωρών των συλλογικών συμβάσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για τις ερωτήσεις σας. Θα δώσω τώρα το λόγο στους προσκεκλημένους μας. Πρώτον ο κύριος Χαράκα και μετά η κυρία Πεκόναν για να απαντήσουν τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και για τις καλές και, εκτετα... και γενικές έτσι, ευρύ, ευρέως ενδιαφέροντος ερωτήσεις. Είμαι και εγώ βουλευτής και καταλαβαίνω ότι χρειαζόμαστε συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, αλλά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, που να καταλάβετε, ότι δεν έχουμε νέα επιτροπή ακόμα, άρα περιμένουμε να ξεκινήσουν οι πρωτοβουλίες της ε, νέας πρόεδρου της Επιτροπής. Δείτε όμως και την άλλη πλευρά του νομίσματος μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα την υφιστάμενη κατάσταση, ούτω ώστε αντί να μπαίνουμε σε θέματα νομοθετικής διατύπωσης των κειμένων, μπορούμε να συζητήσουμε εκτενέστερα στρατηγικές προσεγγίσεις για την, το πρόγραμμα εργασίας και την ημερήσια διάταξη της Επιτροπής και για το αντίστοιχο του Συμβουλίου. Ο κύριος και ρώτησε τι μέτρα θα εφαρμόσουμε για να περάσουμε με δίκαιο τρόπο στην ε, επί, στην, σε μια Ευρώπη που θα είναι ουδέτερη κλιματικά. Στη Γερμανία έχετε μια ε, επιτροπή ανάλυσης των δομών Είναι σημαντικό να έχουμε ανα, αναδιανομή, αλλά η αναδιανομή θα μπορεί να είναι εξίσου σημαντικό να, είναι, να, υπά, με την προκατανομή. Δηλαδή να έχει κανείς δίκαιη αντιμετώπιση πριν την μετάβαση. Αυτό προσφέρει μεγαλύτερες ευκαιρίες και λιγότερες απειλές στους πολίτες ε, ε, της ε, Ένωσης. Μία από τις προτεραιότητες ε, μας είναι η συμπερίληψη. Άτομα δηλαδή που έχουν μερική δυνατότητα απασχολησιμότητας, για παράδειγμα άτομα με αναπηρίες και που πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτή την μετάβαση. Προετοιμάζουμε συμπεράσματα του Συμβουλίου για την αύξηση τη συμπεριλήψη στην αγορά εργασία και μιλούμε για όλους, νέους, ηλικιωμένους, μετανάστες και άτομα που έχουν περιορισμένη ικανότητα απασχολησιμότητας. Και εδώ υπάρχει μεγάλη, ε, υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Η κυρία Μπίσοφ αναφέρθηκε και σωστά στην ελευθερία των συλλογικών συμβάσεων και τη γενικότερη, η γενικότερη συζήτηση ωστόσο του Εργατική της εργατικής νομοθεσίας είναι κομμάτι και του κοινωνικού διαλόγου και η Προεδρία παράσχει ένα πλαίσιο για να μπορέσει να γίνει συζήτηση των διαφόρων πτυχών της εργατικής νομοθεσίας. Ε, ε, η κινητικότητα των εργαζομένων τώρα και οι ρυθμίσεις του και οι σχετικές ρυθμίσεις του Παγκόσμιου Γραφείου ε, Εργασίας. Πιστεύω ότι αυτό μπορεί να γίνει χωρίς νομοθετική παρέμβαση με καλύτερη προστασία απλώς των δικαιωμάτων εργαζομένων. Αυτά είναι τα βασικά μου σχόλια. Θα επανέλθω αν θέλετε και μεταγενέστερα. Κυρία Υπουργέ. Ευχαριστώ. Και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους ερωτώντες για τα πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα που έθεσαν. Πολλοί από εσά σχολιάσετε πράγματα που και εγώ σκέφτομαι, ιδίως Άκουσα τις παρεμβάσεις της ε, Προέδρου, της νέας Προέδρου της Επιτροπής και έχει υπογραμμίσει πολλές φορές τη σημασία των δράσεων ευημερία και κοινωνικά ζητήματα, τονίζοντας ότι αυτά θα είναι στον πυρήνα των δράσεών της. Πιστεύω ότι αυτά ταιριάζουν πολύ με αυτό που εμείς έχουμε στο μυαλό μας, αυτή την οικονομία της ευημερίας. Δηλαδή την ιδέα ότι ο στόχος της δράσης των πολιτικών είναι να είναι καλά οι άνθρωποι, όχι να είναι καλά η οικονομία μόνο. Αυτό αποτελεί και τη βάση μιας κοινωνίας ισότητας. Είναι σημαντικό η ευρωπαϊκή, το ευρωπαϊκό εξάμεινο να λειτουργεί σωστά στο πλαίσιο αυτό και να έχει να συμπεριλάβει και ένα κοινωνικό πυλώνα, μια κοινωνική διάσταση. Θα ήθελα να ακούσω από την επόμενη επιτροπή, τα μέλη της επόμενης επιτροπής, τι συγκεκριμένα μέτρα θα λάβουν σχετικά και θα υποστηρίξω το στόχο της επιτροπής για τα άτομα με τροτότητες, ούτως ώστε να έχουμε μια πραγματικά Ευρώπη της ευημερίας. Η κυρία Βαντελέιεν μίλησε για, και για ειδικά ζητήματα, την ασφάλεια των παιδιών, την ασφάλεια... Θα ήθελα να ξέρω τι εννοεί με αυτό. Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης είναι καθολικό. Όλοι έχουν πρόσβαση στην ευημερία, την κοινωνική ασφάλιση και την εκπαίδευση. Αυτό είναι ένα καλό μοντέλο για μας, το οποίο συστήνω και για άλλους. Σε ό,τι αφορά τώρα την βελτίωση της κοινωνικής διάστασης στην Ευρώπη και τον πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, κάτι που πολλοί ομιλητές σχολίασαν, Ο στόχος μου είναι να βελτιώσουμε τις στρατηγικές μας ώστε η ευημερία της Ευρώπης να ξεκινήσει, να, να προχωρήσει και στο κοινωνικό τομέα. Αυτό το ξεκινούμε στο Συμβούλιο, το ξεκινήσαμε στο Συμβούλιο στην συνάντησή μας στις 8 Ιουλίου με θετικά αποτελέσματα. Ο στόχος μας είναι να έχουμε συμπεράσματα του Συμβουλίου που θα υιοθετηθούν τον Οκτώβριο και για την ισότητα, για την ισότητα να σας πω, και για την, ε, ασφα... αυτά για την, για την ισότητα, για την ασφάλεια. Τα συμπεράσματα θα υιοθετηθούν τον Δεκέμβριο. Θέλουμε να, με τον τρόπο αυτό να εντάξουμε την ευημερία σε όλες τις διαστάσεις πολιτικής. και να κάνουμε και μια σωστή αξιολόγηση αντικτύπου των πολιτικών της Ένωσης. Αυτό ιδίω για τι ευάλωτε κατηγορίες πολιτών, ηλικιωμένοι άτομα με αναπηρίε. και πώ μπορούμε να δώσουμε απαντήσει στα στα άτομα αυτά όταν δεν έχουμε ολοκληρωμένες απαντήσεις πολιτικής. Ο στόχος μας πρέπει να είναι απτά αποτελέσματα στην κοινωνική πολιτική, στην πολιτική υγείας, στην πολιτική κοινωνικής ασφάλισης. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα αυτά είναι αρμοδιότητες των κρατών μελών και είμαστε βέβαιοι ότι τα κράτη-μέλη θα δώσουν έμφαση στην πλήρη προστασία των δικαιωμάτων όλων των ατόμων αυτών, ξεκινώντας πάνω κάτω από την ίδια, από το ίδιο επίπεδο. Ξέρουμε ότι τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στα κράτη-μέλη περνούν συνεχώς από ε, αλλαγές. Ε, οι δυνατότητες της να αναπτύξει ένα ενιαίο σύστημα είναι πολύ περιορισμένες. Ωστόσο, οι, οι ειδικέ ομάδες, η αντιμετώπιση δηλαδή των ειδικών ομάδων είναι θέματα όπως οι ηλικιωμένοι, ε, μετανάστες κλπ. Είναι θέματα που θα συμπεριληφθούν στις συζητήσεις του Συμβουλίου. Είναι σημαντικό να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των πολιτών με δίκαιο και ισότιμο τρόπο. Στη δύσκολη κατάσταση που έχει δημιουργήσει και το Brexit στα πλαίσια αυτά. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύθηκε μονομερώς να προστατεύσει τα κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης και μετά το Brexit. Ελπίζω ότι το ίδιο θα πράξει και η Μεγάλη Βρετανία για τους πολίτες της Ένωσης. Για τα άτομα με αναπηρίες τώρα. Είναι σημαντικό όλα τα άτομα που έχουν κάποιους κινητικούς ή άλλους περιορισμούς να μπορούν να μετάσχουν στην οικονομία της ευημερίας όσο καλύτερα γίνεται. Θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πόρος και όχι ως βάρος στην κοινωνία. Και νομίζω ότι μπορούν να συμβάλλουν με σημαντικό τρόπο ε, και εδώ η Ένωση μπορεί να συμβάλλει με σημαντικό τρόπο στην παροχή δυνατοτήτων για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της αγοράς εργασίας. Υπάρχουν οδηγίες που λένε ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίε πρέπει να είναι προσβάσιμες στην αγορά σε όλους. Ωστόσο υπάρχουν ακόμα περιορισμοί στην πρόσβαση και αυτό θα το συζητήσουμε στο Συμβούλιο στις 24 Οκτωβρίου. Κλείνοντας, για το σύστημα κοινωνική ασφάλισης της Φιλανδίας δύο λόγια. Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι το σύστημά μα έχει δώσει αρκετά καλά αποτελέσματα, ιδίω. για την εξασφάλιση της ευημερία των πολιτών και την καταπολέμηση των αισιοτήτων. Ωστόσο πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι τα συστήματα κοινωνικής ευημερία ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες και καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες και περιπτώσεις. Άρα τα πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε πιο προσεκτικά Όλοι χρειαζόμαστε, όλοι αισθανόμαστε την ανάγκη μεταρρύθμιση των συστημάτων κοινωνική ασφάλιση στι χώρε μα. Ο στόχο μα όμω θα πρέπει να είναι να ε, προσφέρουμε κάποιες βασικές ε, βασικά, βασικά στοιχεία ισότητα σε όλους. είπε είναι ένα σπίτι, μια αιστεία. Είναι σημαντικό, στη Φιλανδία για παράδειγμα έχουμε θέσει ως προτεραιότητα να μην υπάρχουν άστεγοι. Η ψηφιοποίηση για παράδειγμα προσφέρει πολλές δυνατότητες για μια κοινωνική ανάπτυξη που εξασφαλίζει ανάπτυξη και ευημερία. Ταυτόχρονα είναι σημαντικό να προσφέρουμε σε όλους μία ουσιαστική δυνατότητα συμπερίληψης και να περιορίζουμε τον κίνδυνο περαιτέρω αποκλεισμού. Ο στόχος μας, επαναλαμβάνω, είναι να παράσχουμε ευημερία στους πολίτες με πιο αποτελεσματικό και γρήγορο τρόπο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Προχωράμε στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι πάνω από 20 από εσά θέλουν να συμμετάσχουν στη συζήτηση και να θέσουν ερωτήσεις στους προσκεκλημένους μας. Ε, αρκετοί λοιπόν. Ίσως να ζητήσουν ακόμα περισσότερο το λόγο κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Γι' αυτό σύντομα θα αναφέρω τον κατάλογο και κατόπιν θα πρέπει να θέσουμε κανόνες. Madam Fransen, Mr. Kanev, Madam Sander, Madam Galvez, Madam Holmes, Madam Gualmini, uh, Madam Saliba, Madam Brunet, uh, Madam Salani, Madam Lenoir, Madam Vedren, uh, Madam Donat, Mr. Kanes.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 Παρακαλώ. Ωραία. Θα ακολουθήσουμε λοιπόν τους εξής κανόνες. Θα ακολουθήσουμε τις πολιτικές ομάδες, δηλαδή μία πολιτική ομάδα μετά την άλλη κάθε φορά. και νομίζω ότι ήδη είδαμε πόσο δύσκολο είναι να τηρείτε το χρόνο ομιλία σας. Με την εξαίρεση του κυρίου Βίλουμσεν, τον οποίο θα ήθελα να συγχαρώ, όλοι οι άλλοι ξεπέρασαν τα δύο λεπτά. Και έχουμε μεγάλο αριθμό μιλητών. Προτείνω λοιπόν 1,5 λεπτό ο καθένας. Συμφωνείτε? Ωραία. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ να τηρήσετε το χρόνο ομιλίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάμε λοιπόν με την κυρία Σκιτσέταλ. Παρακαλώ. Και είναι παρούσα? Όχι. Σίντι Φράνσεν. Και επόμενη μιλήτρια, κυρία Καλβές, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους υπουργούς που μας παρουσίασαν τις προτεραιότητες της Φιλανδικής Προεδρίας. Δύο ερωτήσεις έχω σχετικά με το Brexit. Το Βέλγιο ε, φαίνεται ότι θα είναι μια από τις χώρες που θα ε, νιώσουν περισσότερο τον αντίκτυπο. Διακυβεύονται 42.000 θέσεις εργασίας. Συμφωνείτε με μια ευελιξία στο Ταμείο ε, Παγκοσμιοποίησης ώστε να στηριχθούν οι εργαζόμενοι που θα χάσουν τη δουλειά τους λόγω του Brexit και επίσης όσον αφορά το χάσμα στις ψηφιακές δεξιότητες. Η Κίνα και, το, και οι Ηνωμένε Πολιτείες ε, αντιπροσωπεύουν το 97% της ψηφιακής οικονομίας, ενώ το 43% των Ευρωπαίων ε, έχουν ελάχιστες έως και μηδαμινές ε, ψηφιακές ε, δεξιότητες. Τι λοιπόν θέλετε να κάνετε για να στηρίξετε τα δικαιώματα των εργαζομένων στο θέμα αυτό. Αυτές είναι οι δύο ερωτήσεις μας. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λίνα Καλβές, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας παρακαλώ η κυρία του Μαντζεντετουπνέη να ετοιμάζεται. Σας ευχαριστώ πολύ για τις εισηγήσεις σας. Ε, σας εύχομαι κάθε επιτυχία ε, κατά τη διάρκεια της Φιλανδικής Προεδρίας. Ε, είπατε, αναφέρατε την οικονομία της ευημερίας, είπατε ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της αηφόρου ανάπτυξης. Ωστόσο, η κατεύθυνση της πολιτικής οικονομίας, της οικονομική πολιτικής τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει σε αύξηση των ε, ανισοτήτων ε, και θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Η ανάλυση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ε, οδηγεί και σε υποδείξεις για το τι θα πρέπει να κάνει κάθε χώρα. Αλλά η ανάλυση αυτή βασίζεται και σε κάποιες ε, υποθέσεις που δεν στηρίζονται πάντα από δεδομένα. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω. Μπορείτε να φροντίσετε παρακαλώ ο νέος ε, ευρωπαϊκός πυλώνας ε, κοινωνικών δικαιωμάτων να ενσωματωθεί σωστά στο ευρωπαϊκό εξάμεινο, διότι μόνο 14 από τα 20 ε, σημεία δεν συνδέονται 14 από τα 20 σημεία του πίνακα αποτελεσμάτων δεν συνδέονται με δείκτες, ενώ τα υπόλοιπα 6 μόνο εν μέρη. Ε, η επόμενη ομιλήτρια, εκτός μικροφώνου. Les ministres, merci pour votre présence. Nous avons beaucoup parlé euh, de l'enjeu de l'énorme décalage. Ευχαριστώ πρόεδρε που ήσασταν εδώ. Υπάρχουν σοβαρές αποκλίσεις μεταξύ των στόχων και της αγοράς εργασίας. Θέλω να σταθώ στους νέους και 14 εκατομμύρια άτομα που δεν, πάνω από 1 εκατομμύριο στην Γαλλία που δεν είναι ούτε σε εκπαίδευση ούτε σε δουλειά. Γι' αυτό το κομμάτι του πληθυσμού τι μέτρα θα λάβετε στο πρόγραμμα της φιλανδικής Προεδρίας μιλάτε για ένα μοντέλο του σούπερ πανεπιστημίου. Πολύ ενδιαφέρον. Σκέφτεστε να περιλάβετε, ας πούμε, για παράδειγμα και νέους εργαζόμενους για μόνιμη επανακατάρτιση. Η κυρία Φίλιπς έχει το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην Προεδρία σας. Η Φιλανδία έχει θέσει πολύ φιλόδοξο στόχο να είναι ουδέτερη ως προς το διοξίδιο του άνθρακα μέχρι το 2030 και σίγουρα η ηγείται είναι πρωτοπόρος στον τομέα αυτό. Ε, είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτή η μετάβαση. Όσον αφορά την απασχόληση, Τι έχετε προτείνει για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ε, για να διασφαλίσετε μια πιο δίκαιη μετάβαση. Ε, σας ευχαριστώ πολύ, ο Σκόρτιν, και η κυρία Σαΐμπη να ετοιμάζεται. Καλημέρα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την επισκόπηση ε, της Προεδρίας σας. Εγώ απογοητεύτηκα με τα όσα άκουσα. Πολλά κλισέ ακούσαμε, πολύ λίγα συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ θα ήθελα να ξέρω συγκεκριμένα τι θα κάνετε για τους ε, νέους ανθρώπους και στον κοινωνικό τομέα. Μόνο μία φορά άκουσα τη λέξη «οικογένεια». Είπατε κοινωνικές υπηρεσίες για όλες τις ε, οικογένειες. Για μένα που προέρχομαι από το, από το ε, πολιτικό κόμμα των οικογενειών της Γερμανίας, ε, αυτό μου κακοφαίνεται. Πιστεύω ότι οι οικογένειες θα στηρίξουν την Ευρώπη, αλλά πολλές οικογένειες στην Ευρώπη περνάνε πολύ δύσκολα. Και η κυρία Ούρσουλα Φονταλάιεν αναφέρθηκε στο θέμα αυτό. Θέλουμε να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των οικογενειών, να ενισχύσουμε τις οικογένειες, διότι εκεί βρίσκονται οι ρίζες της δημοκρατίας μας. Και αυτό θα καθορίσει την ε, συνύπαρξή μας στην Ευρώπη. Πολύ απογοητευμένος είμαι λοιπόν. Σας εύχομαι καλή Προεδρία και ελπίζω από κοινού να μπορέσουμε να βρούμε το δρόμο προς μια Ευρώπη των οικογενειών, Ευρώπη της οικογένειας. Ευχαριστώ. Η κυρία Σαϊπή. Και ο κύριος Νικολάου να ετοιμάζεται παρακαλώ. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Μιλήσατε για το θέμα της στέγης, που είναι βάση οποιασδήποτε προσπάθειας ε, αξιοπρεπούς ζωής και κοινωνικής ένταξης. Και σωστά, κύριε Υπουργέ, μιλήσατε για τους άστεγους. Η Φιλανδία θεωρείται ως ένα μοντέλο για την πολιτική στέγαση που έχει στόχο να επιτρέψει σε άστεγους να μπορέσουν να αποκτήσουν στέγη, όχι να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του, της έλλειψης στέγης με προσωρινή στέγη. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και στην ε, διαπίστωση που έγινε πρόσφατα ότι το ποσοστό του οικογενειακού εισοδήματος για τον νίκη αυξάνεται όλο και περισσότερο στην Ευρώπη. Υπάρχουν χώρες, η Ολλανδία για παράδειγμα, όπου υπάρχει μια βολοταριστική πολιτική ε, οικοδόμησης εργατικών κατοικιών, μαζικής οικοδόμησης εργατικών κατοικιών, που ε, ε, υφίσταται κυρώσεις από την Κομισιόν, η οποία αναφέρει ότι στέγη η πολιτική στέγης πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες ε, του ανταγωνισμού και ότι δεν είναι ε, κρατική πολιτική. Άρα ότι δημιουργούσε η κατασκευή εργατικών κατοικιών θέμει τον ανταγωνισμό σε σχέση με την ιδιωτική αγορά. Αυτό επιβαρύνει την κρίση της στέγης σε όλη την Ευρώπη. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Ο κύριος Νικολάου και ο κύριος Κάνευ κατόπιν. Όπως και στις υπόλοιπε χώρε τη Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυστηρότητα ε, εφαρμόστηκαν και εξειδικεύτηκαν οι νομοθεσίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό την προηγούμενη οκταετία έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Μείον 20% ε, στο μέσο μισθό, μείον 35% στο μέσο μισθό για την ελαστική απασχόληση, αύξηση τη ελαστική απασχόληση, διατήρηση πολύ υψηλών. Ε, πολύ ψηλή ανεργία, ιδιαίτερα για του νέου, όπου φτάνει και είναι στα 40% διάλυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων σχεδόν σε όλου του κλάδου τη οικονομία. Αποδεικνύεται ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία, ο ευρωπαϊκό πυλώνα δικαιωμάτων, η κινητικότητα δεν έρχεται να αντιστρέψει αυτή την πραγματικότητα, αλλά στην πραγματικότητα να δράσει συμπληρωματικά σε αυτήν. Εγγυάται δηλαδή ένα πολύ χαμηλό, ελάχιστο επίπεδο διαβίωση, κάτω και από αυτά τα όρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται οι όροι έτσι ώστε να καθιζάνουν συνολικά το επίπεδο των δικαιωμάτων των μισθών προ τα εκεί ακόμη και σε, ε, μετά από γενικευμένη κατακραυγή για τις καταγγελίες για τους όρους εργασίας σε μεγάλα μονοπόλια, όπως για παράδειγμα στην Amazon στη Βρετανία ή ε, τις προηγούμενες μέρες που είχαμε ένα μεγάλο σεισμό στην Ελλάδα όπου οι εργαζόμενοι των μεγάλων εταιριών αναγκάστηκαν να μπουν μέσα να δουλέψουν μετά το σεισμό, τι κάνουν τα κράτη-μέλη. Υιοθετούν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ιταλία, στο Βέλγιο, στη Σουηδία, στη Βρετανία νομοθεσία η οποία περιορίζει τη δυνατότητα κινητοποίηση των εργαζομένων, περιορίζει την ικανότητα να παίρνουν απόφαση για απεργιακέ κινητοποιήσει. Οι ίδιε οι ελεγκτικέ αρχέ των κρατών είναι ξεχαρβαλωμένε και τώρα αποθέτουμε τι, μια, σε μια ευρωπαϊκή ε, αρχή εργασία να έρθει να διαπιστώσει και να προσανατολίσει σε τι. Να προσανατολίσει ότι χρειάζεται να μειωθούν οι αποδοχέ, ότι χρειάζεται να αυξηθεί η ελαστική απασχόληση, ότι χρειάζεται να απαγορευτεί η οργάνωση τη εργατική τάξη στου χώρου δουλειά, να αφηθούν οι εργαζόμενοι έκθετοι στου εργοδότε. Θα θέλαμε μια τοποθέτηση της Φιλανδικής Προεδρίας για αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Mr. Ο κύριος Κάνιεφ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Και η κυρία Ελίσσα Χόλμς, παρακαλώ, προετοιμαστείτε. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι Υπουργοί, θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Όλοι πιστεύω ομόφωνα και ευρέως υποστηρίζουμε σε αυτό το κοινοβούλιο ότι υπάρχει ανάγκη για μια πιο δραστήρια κλιματική πολιτική. Επίσης πιστεύω υπάρχει ευρεία συνένεση για μια σωστή μετάβαση, ειδικότερα για τις βιομηχανικές περιοχές, για τις βασικές ε, περιοχές που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην ε, παραγωγή άνθρακα. Εγώ ως Βούλγαρος ε, ε, ζω σε μετάβαση εδώ και 30 χρόνια. Και ξέρω ότι καμία μετάβαση δεν είναι τόσο δίκαιη όσο τη φανταζόμαστε αρχικά. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω κατά την άποψή σας ποιο απτά μέτρα για την αγορά εργασίας, ε, ενέργειας ε, στον τομέα της εξόρυξης για αυτή τη μεταβατική περίοδο. Για να έχουμε μια δίκαιη μετάβαση. Πιστεύω η Φιλανδία έχει αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα στο παρελθόν, οπότε έχετε και εσείς προσωπική εμπειρία. Ευχαριστώ κυρία Άισα Χόλμς και η κυρία Σαλάνη. Παρακαλώ, ετοιμαστείτε. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστούμε τους κύριους Υπουργούς που βρέθηκαν εδώ σήμερα για να μας ε, κάνουν αυτή την ενημέρωση για θέματα απασχόλησης και κοινωνικών θεμάτων. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά την απασχόληση και η δεύτερη τα κοινωνικά θέματα περισσότερο. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα οι νέοι στην Ευρώπη και η απασχόλησή τους. Η σημερινή γενιά είναι πολύ δικευμένη, πολύ καταρτισμένη, αλλά αντιμετωπίζει το κενό δυνατοτήτων. ελάχιστε θέσει εργασία, αβέβαιη εργασία, χαμηλέ, αμοιβέ χωρίς ε, καμία προοπτική και χωρίς καμία όρεξη να ξεκινήσει κανεί μια σταδιοδρομία γιατί δεν έχει δυνατότητε. Τι μέτρα λοιπόν προβλέπετε εσείς ε, για να αντιμετωπιστεί η ενεργεία των νέων και για να βρεθούν ε, αξιοπρεπείς δουλειές για τους νέους. Δεύτερη ερώτηση, τι γίνεται με τους ανέργους, με τους συγγνώμη, άστεγους ε, που δεν έχουν πάρα πολλά δικαιώματα, στερούνται πολλών δικαιωμάτων. Η Φιλανδία είναι πρωτοπόρος όσον αφορά το Housing First. Εσείς ως Προεδρία θα διασφαλίσετε το δικαίωμα των πολιτών να έχουν μια αξιοπρεπή ε, κατοικία ή συνθήκες διαβίωσης. Ευχαριστώ. Κυρία Σαλάνη, έχετε το λόγο. Και κυρία Λίζη, παρακαλώ, ετοιμαστείτε. Θα ήθελα να μιλήσω ειδικά αυτή τη φορά. Σας ευχαριστώ, Προεδρή, κυρία Πρόεδρε, για το λόγο και ευχαριστώ τους υπουργούς που είναι παρόντες. Ε, ακούσαμε τα μελλοντικά σας σχέδια, ακούσαμε και τις απαντήσεις που δώσατε στις ερωτήσεις. Βρίσκω ότι είναι πολύ καλή ιδέα να κοιτάξει κανείς την καρδαρόπα του, ε, την τουλάπα του, προτού πάει να αγοράσει ρούχα. Ε, να μην ε, ψάχνουμε για νέα ε, πράγματα προτού εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας. Έχουμε υποσχεθεί πολλά στους ε, ψηφοφόρους μας αυτές τις εκλογές και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ένας φορέας που ενισχύει τους πολίτες. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω η Φιλανδική Προεδρία πώς σκέφτεται να διασφαλίσει ότι οι προτάσεις που υποβάλλονται δεν θα επιδεινώσουν τις συνθήκες για τους εργαζομένους. Δεύτερον, είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, η Φιλανδική Προεδρία να ασχοληθεί με φαινόμενα που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ζήνη, έχετε το λόγο και κυρία Ζελέσκα, παρακαλώ ετοιμαστείτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ του υπουργού από την Φιλανδία ε, που θα δείξουν τόσο μεγάλη αφοσίωση στον τομέα τη απασχόληση. Ένα από του πυλώνε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Φιλανδία αντιπροσωπεύεται από τη μετάβαση προ μια ουδέτερη κλιματικά κοινωνία. Συχνά μας υπενθυμίζουν ε, έννοιες όπως την ε, παγκόσμια ανακατανομή της εργασίας, το σχηματισμό της εργασίας, την ψηφιοποίηση ε, με επικοδομητικές προοπτικές. Η Φιλανδική Προεδρία σκοπεύει να βοηθήσει να εξισορροπηθεί η μετάβαση και να προστατευτούν οι εργαζόμενοι στους παραδοσιακούς όπως ονομάζονται τομεί, χωρίς να αφήσουμε πίσω κανέναν. Με ποια εργαλεία και με ποιους πόρους ε, σκοπεύετε να συνοδέψετε την μετασχηματισμό αυτό των ευρωπαϊκών λαών καθώς θα περνάμε από τη σημερινή οικονομία στην ουδέτερη κλιματικά οικονομία. Ποια βήματα, με ποια βήματα θα γίνει η μετάβαση αυτή. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενδέχεται να μην έχουν τα επαρκή εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τέτοιου επανάσταση πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε τις κρίσεις απασχόλησης που θα έχουμε μετά από τεχνολογικές μετασχηματισμούς στις κλασικές επιχειρήσεις σε παγκόσμιο ε, πλαίσιο έχουν υπάρξει τέτοιες ε, ανισορροπίες οικονομικές ε, κατά τη μετάβαση ορισμένων οικονομιών σε νέους τομείς. Μετά όσον αφορά την κινητικότητα των εργαζομένων τι γίνεται ε, σε αυτό, σε συνδυασμό με τη ε, διάφορα κλιματικά θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό εξάμεινο. Ευχαριστούμε κύριε Ζαλεύσκα. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Κύριε Πάτσαν, ετοιμαστείτε. E, e, Κυρία Πρόεδρε, ε, υπόθηκε ότι στην ουσία η Φιλανδική Προεδρία ε, θα διαρκέσει τρεις μήνες. Όλα εξαρτώνται από το πότε θα ε, συσταθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ερώτηση. Τι πιστεύετε για τον προϋπολογισμό που έχει υποβάλει η παρούσα ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον έχει απορρίψει πώς βλέπετε τις δυνατότητες για περαιτέρω διαπραγματεύσει πάνω στον προϋπολογισμό αυτών. Ε, άλλο θέμα, επανάσταση 4.0, ε, τεχνολογική επανάσταση. Ο κύριος Υπουργός ε, μίλησε για τις νέες δεξιότητες και είπε ότι η εκπαίδευση μέχρι στιγμής δεν ήταν αρκετά αποτελεσματική. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι τι λύσεις προτείνετε ώστε οι ενήλικες να έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να ανταποκριθούν στην Επανάσταση 4.0. Η στρατηγική 2020 προέβλεπε να υπάρχουν περισσότεροι με επιτυχία πανεπιστημίων. Αλλά ξεχάστηκαν οι ενδιάμεση και τελευταία ερώτηση σχετικά με την απασχόληση. Ε, ναι, κοιτώ το χρόνο, έχω κι άλλο χρόνο στη διάθεσή μου. Ελέγχω το ρολόι. Συγγνώμη, διακόπτη η πρόεδρος. Ο κύριος Πάτεν και μετά η κυρία Σάντερ μπορεί να ετοιμαστεί. Ευχαριστώ. Έχω δύο ερωτήσεις. Έχω μπερδευτεί με την απάντηση του κυρία, της κυρίας Πεκόνων για την ερώτηση που αφορούσε το Brexit και τα δικαιώματα των πολιτών μετά το Brexit. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προστατεύσει και είπε ότι θα διασφαλίσει τα δικαιώματα των 3,2 εκατομμύριων Ευρωπαίων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εσείς προτι... Ε, υπενήσεστε στην απάντησή σας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει το ίδιο για τους Βρετανούς πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να το ξεκαθαρίσετε παρακαλώ. Δεύτερον, θέλω να σκεφτείτε πιο ε, μυαλα για το Brexit και το πώς συνέβη. Ε, συνέβη για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων ήταν η απεριόριστη ροή οικονομικών μεταναστών προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κόσμος αισθανόταν ότι έχανε τις δουλειές του, ε, μειώθηκαν οι μισθοί, οι τοπικέ κοινότητες αισθανθήκαν ότι δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Έλαβε ε, τεράστιο πλήγμα απόψη κοινωνικών ε, ε, ωφελών η Βρετανική οικονομία. Η κυρία Βαντελέιεν μίλησε στο Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα και είπε ότι ο κόσμος χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη και αναφέρθηκε στην ιδέα ενό κατώτατου μισθού πανευρωπαϊκού, μια ένωσης κεφαλαίου αγορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, μιας ε, εταιρικής φορολογικής βάσης ε, πανευρωπαϊκής και θέλω η Προεδρία να μου πει το εξή. Όπως φαίνεται υπάρχουν βαθιές διαφορές μεταξύ εθνών, μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας για παράδειγμα, μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Συμφωνείτε ότι αυτές οι πολιτικές από πάνω προς τα κάτω τις οποίες ακούμε τόσο πολύ τελικά δεν λειτουργούν. Δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της απόδοσης. Στη... Έχουν δοθεί ένα σωρό λεφτά στην Ισπανία και ένας στους τρεις είναι άνεργος τα δημοκρατικά κράτη, τα κυρίαρχα κράτη είναι το καλύτερο μέλος, ε, μέρος για να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Παρακαλούμε να ενθαρρύνετε περισσότερο τα κράτη-μέλη αντί για τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Uh, κυρία Αν Σάντερ και κυρία Γκουαλμίνη, παρακαλώ ετοιμαστείτε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, λοιπόν, κάνει ζέστη σήμερα στις Βρυξέλλες και παντού στην Ευρώπη. Όχι εδώ σε αυτή την αίθουσα, ευτυχώ. Όταν κάνει ζέστη, συχνά λοιπόν εκδηλώνονται πυρκαγιέ παντού στην Ευρώπη. Και σήμερα περισσότερο από ότι είναι φυσιολογικό. Παραπάνω λοιπόν από ό,τι συνηθίζεται, χρειαζόμαστε πυροσβέστες και εθελοντέ πυροσβέστε, ειδικότερα στις αγροτικές περιοχές. Αυτοί είναι οι πρώτοι που παρέχουν βοήθεια στους συμπολίτες μας. Το σύστημα αυτό των εθελοντών πυροσβεστών υπάρχει κίνδυνος ε, να υποβαθμιστεί λόγω μιας απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που θεωρεί ότι ο χρόνος διαθεσιμότητας αυτών των εθελοντών πυροσβεστών μπορεί να θεωρηθεί χρόνος εργασίας. Και εκεί η οδηγία που αφορά τους χρόνους εργασίας ε, μπορεί να υπονομεύσει αυτό το σύστημα των εθελοντών πυροσβεστών. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε την άποψή σας επί του θέματος. Πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσατε εσείς να μας βοηθήσετε, να βοηθήσετε τις χώρες που τα διάφορα κράτη-μέλη για να κάνουμε μία πρόταση, ούτως ώστε να προσαρμόσουμε ε, τη λύση και, ώστε να διατηρηθεί αυτό το σύστημα βοήθειας παντού στα κράτη-μέλη μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ελιζαμπέτα Γκουελμίνη, έχετε το λόγο. Και παρακαλώ να ετοιμάζετε η κυρία Λενουάρ. Ναι, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έχω μια γενική παρατήρηση και δυο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Η παρατήρηση Απίλασα γενικά το γενικό πλαίσιο που μας ε, περιγράψατε και οι δύο, που μας και γραφήσατε κοινωνικές ε, ε, συνθήκες καλές, η κοινωνική ευημερία αποτελούν προϋπόθεση της οικονομικής ανάπτυξης. Η οικονομική ανάπτυξη δηλαδή πρέπει να συνοδεύεται από ένα κράτος ευημερίας και από την κοινωνική προστασία. Και φυσικά, όπως είπε, μας είπε η κυρία Πεκόναν, η ευτυχία δεν είναι για τους λίγους, αλλά για τους πολλούς. Ας το θυμόμαστε λοιπόν. Ε, πρώτε Πρώτη μου ερώτηση λοιπόν, κυρία Πεκόναν, αναφέρατε του ηλικιωμένου. Θα μπορούσατε να είστε λίγο πιο ακριβείς. Μιλήσαμε πολύ για την εγγύηση για τα παιδιά, αλλά ξέρετε η Ευρώπη γυράσκει διαρκώς. Μπορείτε να μου πείτε λοιπόν τι προτίθεστε να προωθήσετε όσον αφορά την ενεργό γύρανση και για τους ηλικιωμένους. Η δεύτερη μου ερώτηση έχει να κάνει με την ισότητα των φύλων. Όπως ξέρετε υπάρχουν ήδη αρκετές συστάσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την μείωση του μισθολογικού χάσματος ε, και για την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματική ζωής. Μπορείτε να μας δώσετε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Λενουάρ. Έχετε το λόγο. Και παρακαλώ κυρία Ζαμπέλη αν προετοιμαστείτε. Ευχαριστώ. Κυρία και κύριε Υπουργέ, καταρχάς να τονίσω πόσο εκτιμώ την προσπάθειά σας για μια Ευρώπη περισσότερο ανοιχτή και συμπεριληπτική, ιδίω τα άτομα με αναπηρίες. Συχνά τα άτομα με αναπηρίες δυσκολεύονται να μπουν στην αγορά εργασίας, όπως και άτομα που έχουν υποστεί μεγάλη θεραπεία που έχει φυσιο, φυσιοσωματικές επιπτώσεις χημειοθεραπεία για παράδειγμα. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ε, επανένταξη στην αγορά εργασίας μετά από ένα καρκίνο ή την Ευρωπαϊκή Δομή επιστροφή της μετά από ασθένεια ατύχημα. Το Συμβούλιο έχει προβλέψει να λάβει υπόψη στον τομέα αυτό τη δουλειά που έχει ήδη γίνει σχετικά και τι μέτρα θα υιοθετήσει για να προσθέσει ευρωπαϊκή προστιθεμένη αξία. Χαίρο που έμαθα ότι η Φιλανδική Προεδρία θα οργανώσει μία διάσκεψη για τον επαγγελματικό καρκίνο στο, Περσί, στο Ελσίνκι. Ωστόσο, δυστυχώς αυτό γίνεται κατά τη διάρκεια μιας ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Ζαμπέλη και Ροντινέλη κατόπιν. Κοίτα, κοίτα. E Καλημέρα, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Φιλανδική Προεδρία και το Συμβούλιο για την παρουσίαση του πολιτικού προγράμματος εργασίας της κατά το επόμενο εξάμεινο. Δεν είδα μεταξύ των προτεραιοτήτων της ένα σημαντικό θέμα τους ανηλίκους, ιδίως εκείνους που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση. Σας τονίζω την περίπτωση μιας, μια περίπτωση που έχει, ε, που έχει δημιουργήσει σοβαρή ανησυχία σε όλη την, ε, την Ιταλία, στην περιοχή της ε, Μύρια Ρωμάνια, στο Μπιμπιάνο, με, με, και έχει δημιουργήσει σειρά ζητημάτων ε, παρέμβασης κράτους και επαγγελματιών για να ζητήσουν από τα παιδιά να περιγράψουν το τι έχουν υποστεί ε, για να τα ε, έχουν υποστεί με, με, το επιχείρημα ότι έχουν υποστεί σοβαρές ε, παραβιάσεις των προσωπικών τους δικαιωμάτων που δεν έχει συμβεί με στόχο να τους πάρουν από οικογένεια, την οικογένειά τους και να τους δώσουν σε άλλες, ε, σε άλλες οικογένειες. Αυτό έχει ένα τεράστιο ζήτημα χωρίς καμία, κανένα προηγούμενο στην Ιταλία. Θα υποβάλω μια προφορική ερώτηση που και ένα ευρωπαϊκό αίτημα επιρροής. Είμαι μητέρα και φοβάμαι, οργίζομαι για αυτό που συμβαίνει αν συμβεί κάτι τέτοιο σε εμά. Γι' αυτό ζητώ από την Φιλανδική Προεδρία να συμπεριλάβει μεταξύ των προτεραιοτήτων της κυρία Ζαμπέλη. Δεν έχουμε χρόνο γι' αυτό. Δεν μπορώ να σας επιτρέψω να κάνετε κάτι. Αυτό είναι άδικο προς όλους τους άλλους συναδέλφους. Ροντινέλη. Και η κυρία Βεντρέν κατόπιν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ τους υπουργούς για την παρουσίαση της Φιλανδικής Προεδρίας, ιδίως σε ό,τι αφορά την οικονομία της ευημερίας. Δύο ερωτήσεις θέλω να θέσω με βάση και αυτά που ακούστηκαν μετά τις παρεμβάσεις των συντονιστών αλλά που δεν απαντήσατε εσείς. Και θέλουμε την άποψή σας για αυτά τα δύο ζητήματα. Πρώτον, βγαίνουμε από χρόνια λιτότητας που οδήγησαν ολόκληρες χώρες και περιφέρειες ε, της Ένωσης να ε, περικόψουν τις ε, κοινωνικές δαπάνες για πολλούς πολίτες. Ε, τι θα κάνετε για την ενίσχυση του κοινωνικού πυλώνα. Η αγορά εργασία, το δεύτερο θέμα, δεν έχει δώσει πλονεκτήματα, δεν έχει δώσει κέρδη στους πολίτες σε ό,τι αφορά την κοινωνική πολιτική. Θα ήθελα να έχει επίγνωση αυτού του γεγονότος η Φιλανδική Προεδρία ε, στρέβλωση του ανταγωνισμού που στηρίζεται στο κοινωνικό ντάμπινγκ από απομάκρυνση δε επιχειρήσεων λόγω χαμηλότερων μισθών σε άλλες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι λύση. Δεν υπάρχει, μη έχοντας άλλο τρόπο να περιοριστεί, να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα χρησιμοποιούμε το το εργασιακό κόστος σαν μόνο εργαλείο μείωσης του κόστους. Θα πρέπει η, Σουηδική, η Φιλανδική Προεδρία να μας απαντήσει πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα του αθέμητου ανταγωνισμού. Βεντρέν. Και κατόπιν ο κύριος Σαλίμπα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ για την παρουσίασή σας εδώ. Συμμεριζόμαστε τις κοινέ φιλοδοξίες σας για την κοινωνική συμπερίληψη. Χαίρομαι γι' αυτό. Μία ερώτηση θέλω να κάνω για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα. Συμφωνείτε με το Κοινοβούλιο για την μείωση του ορίου στις 200 καταργήσεις θέσεων εργασίας ε, ε, σε 6 μήνες και όχι 250 σε 4 μήνες. Δεύτερον, πώς εξετάζεται την ε, λήψη υπόψη του, της κοινωνικής διάστασης της συστάσης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σαλίμπα. Και μετά η κυρία Ντόνατ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ αξιότιμοι Υπουργοί για τις παρουσιάσεις σας και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για την ε, Φιλανδική Προεδρία. Περίπου 25 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 18 ετών ε, έχουν τον κίνδυνο φτώχειας ε, ή κοινωνικού αποκλείσμου και δυστυχώς πρόκειται για έναν φαύλο κύκλο τα παιδιά που είναι φτωχά σήμερα. Αύριο θα γίνουν γονείς που θα κάνουν παιδιά τα οποία επίσης θα διατρέχουν τον κίνδυνο της ένδυας. Η νέα Πρόεδρο τη Κομισιόν πριν μια εβδομάδα δεσμεύτηκε στην πρώτη ομιλία να καταβάλει προσπάθειε για να δημιουργηθεί ε, το σύστημα προστασία των παιδιών ε, Εγγύηση ε, για τα παιδιά. Είναι μια ιδέα που ξεκίνησε το Κοινοβούλιο και το πρόθεσε η δική μου πολιτική οικογένεια, οι Σοσιαλδημοκράτε. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω κατά πόσο η Προεδρία έχει κάποια πρόθεση να υιοθετήσει αυτή την πρωτοβουλία και να κάνει κάτι για αυτήν και πιο σημαντικό ακόμα να την προωθήση στο Συμβούλιο. Και αν το πράξετε αυτό, έχετε ήδη ξεκινήσει συζητήσει με κράτη-μέλη για να δείτε ποιε είναι οι αρχικέ του αντιδράσει. Χρειαζόμαστε να βοηθήσουμε ε, ώστε κάθε παιδί που διατρέχει κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού ή φτώχεια στην Ευρώπη να έχει, αν μη τι άλλο, πρόσβαση σε βασικά δικαιώματα όπω ε, υγειονομική περιθέλψη και παιδεία. Αλλά πάνω απ' όλα χρειαζόμαστε πρώτα απ' όλα όλες τις πολιτικές προσπάθειες από όλες τις πλευρές ώστε να υλοποιηθεί η ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά. Ευχαριστώ κυρία Ντόνερ και ο κύριος Κάρας μπορεί να προετοιμάζεται. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω γκρικά και ζητώ συγγνώμη. Ε, ε, ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, τονίζετε ως Φιλανδική Προεδρία ότι έχετε την προτεραιότητα παροχής ε, ισότητας των φύλων. Κάτι που φυσικά είναι ευπρόσδεκτο. Ήθελα να σας ρωτήσω, από το 1957, από τη συνθήκη της Ρώμης, καθόμαστε και συζητάμε για ίσες αμοιβέ και έκτοτε συνεχίζεται να υπάρχει αυτό το μισθολογικό χάσμα. Δεν υπάρχουν ίσες ευκαιρίες ουσιαστικά τι, πώς θα κάνει τη διαφορά η Φιλανδική Προεδρία, δηλαδή σχεδιάζεται να κάνετε κάποια βήματα ώστε να φύγουμε από αυτό το αδιέξοδο. Επίσης αναφέρατε ότι η Φιλανδική Προεδρία θα ήθελε να ε, εντείνει την κινητικότητα και την πρόσβαση σε υψηλά καταρτισμένους εργαζομένους. Εγώ ήθελα να τονίσω ότι η κινητικότητα των υψηλά καταρτισμένων εργαζομένων σε ορισμένα κράτη-μέλη ουσιαστικά σημαίνει διαρροή εγκεφάλων, brain drain, Εσεί ε, πώ σκοπεύετε να μετριάσετε τι ε, συνέπειε, όπω για παράδειγμα στην υγειονομική περίθαλψη, και τις ορισμένε χώρε ε, είναι δύσκολο πλέον να παρέχει κανεί υπηρεσίε υγειονομική περίθαλψη, γιατί έχουν φύγει οι γιατροί στην Ουγγαρία, α πούμε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όλη μέρα άκουγα την κυρία Βαντελέ να δεσμεύεται για σημαντικά ζητήματα μεταξύ των οποίων να παροτρύνει έναν ευρωπαϊκό ελάχιστο μισθό, μια εγγύηση για το παιδί. Σας άκουσα και εσάς προσεκτικά. Από ό,τι φαίνεται οι δικές σας δεσμεύσεις πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Κάποια στιγμή λοιπόν θα έπρεπε ίσως να συμφωνήσουμε σε κάποιους κοινούς στόχους καταπολέμησης των βασικών προβλημάτων της Ευρώπης που ζητούν και εκείνων που ζητούν να πάμε πίσω και όχι να πάμε μπρος, που δημιουργούν αβεβαιότητες αντί να χτίζουν βεβαιότητες. Θα ήθελα να υπάρχει μια απλή απάντηση λοιπόν που θα δίνει ελπίδα και δέσμευση σε τρει, σε πέντε, σε έξι μήνες, αλλά ε, το ξεκίνημα είναι πάντα σημαντικό σε αυτή την ε, θητεία μας. Δεσμεύεται η Προεδρία μας σας να προωθήσει τον κοινωνικό πυλώνα της Ευρώπης ως εγγύηση για την οικοδόμηση μιας πιο δίκαιης Ευρώπης ε, που έχει στόχο τη βελτίωση των πολιτών της. Η κυρία Ραφαέλα. Ευχαριστώ για τις προσπάθειες που κάνετε. Χαίρομαι που διαβάζω ότι η Φιλανδική Προεδρία πιστεύει ότι δεν μπορεί να χάσει κανένα κομμάτι από το κεφάλαιο του, των πολιτών της ούτε να και, δε... και θέλει να αντιμετωπίσει τον ρατσισμό. Τι μέτρα προτίθεται ωστόσο να λάβει για να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό. Δεύτερη ερώτηση. Οι νέοι χρειάζονται ειδική προσοχή. Στο πρόγραμμά σας είπατε ίσες ευκαιρίες για όλους ανεξάρτητα από την προέλευσή τους. Θα ήθελα να ξέρω τι μέτρα συγκεκριμένα προτείνεται για το σκοπό αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα μια σημαντική ερώτηση. Ξεχάσαμε κάποιον. Υπάρχει κάποιος που ήθελε να πάρει το λόγο ενώ ήθελε να μιλήσει. Όχι, ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα περάσουμε στον δεύτερο γύρο απαντήσεων. Δεν σας ζηλεύω, κύριε και κυρία Υπουργέ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είπατε ότι δεν μας ζηλεύετε. Ε, να μας ζηλεύετε όμως, διότι ήταν πάρα πολύ καλές οι ερωτήσεις που μας θέσατε. Οι ερωτήσεις αυτές δείχνουν βαθιά γνώση ε, και μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε περισσότερο σε βάθος σε θέματα που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου ερωτήσεων. Να μας ζηλεύετε λοιπόν. Είναι μεγάλη μας χαρά να είμαστε εδώ. Τέθηκαν κάποιες ερωτήσεις σχετικά με κάποια ταμεία, σχετικά με τις δεξιότητες, την ανάπτυξη, την προστασία των εργαζομένων. Και έχουμε φυσικά και το Brexit, το θέμα της ημέρας. Είναι κάτι που μας αφορά βαθύτατα. Η εφαρμογή της ελεύθερης κυκλοφορίας ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα σταματήσει αν έχουμε τελικά σκληρό Brexit, Brexit χωρίς συμφωνία. Είχα συζητήσεις με τους συναδέρφους υπουργούς μου σχετικά με την κατάσταση μετά την 1η Νοεμβρίου. Οι συνάδελφοί μου που είναι υπεύθυνοι για τις εξωτερικές σχέσεις ε, λένε ότι ε, έχουν γίνει κατάλληλες προετοιμασίες. Το θέμα αυτό όμως ε, συνδέεται πράγματι με το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης και το Συμβούλιο έχει πάρει θέση στο θέμα αυτό που συμπεριλαμβάνει την αρχική ιδέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θεωρεί ότι ε, ε απότομες αλλαγές στο εμπόριο, για παράδειγμα, μπορούν ε, να οδηγήσουν σε εκταμίευση πόρων. Αυτό λοιπόν θα καλύψει και το Brexit. Αναφέρθηκε η ενεργειακή μετάβαση και πράγματι είναι πολύ επώδυνες οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν από χώρες που χρησιμοποιούν πολλά όρυκτα καύσιμα. Απομένει να δούμε αν ε, η πρόταση της Ursula von der για ένα ταμείο δίκαιης μετάβασης ε, θα εφαρμοστεί. Επίσης, ε, αναφέρθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινό Ταμείο ΣΥΝ. Αυτό είναι κάτι που θα το επιδιώξω στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Είναι σημαντικό να έχουμε ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική και να εφαρμόσουμε τον ε, ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Το Συμβούλιο ήταν ικανοποιημένο με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απλοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας στον κοινωνικό τομέα και να προχωρήσουμε σε περαιτέρω απλούστευση, ε, μεγαλύτερη ευελιξία και αναλογικότητα ε, για τα κράτη-μέλη. Είμαστε διατεθειμένοι να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο γίνεται συντομότερα. Αναφέρθηκε η ψηφιοποίηση. και ίσως θα έπρεπε να αναφέρουμε ότι το Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε πριν δύο εβδομάδες κατέληξε σε συμπεράσματα σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Τονίσαμε τη σημασία των επενδύσεων και του εμπορίου. Έχουμε όμως και ανησυχητικά νέα. Η έλλειψη δεξιοτήτων στον τομέα της ψηφιοποίησης αποτελεί απειλή για την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε ψηφιακές δεξιότητες σε σχεδόν παντού στην αγορά εργασίας. κατά τη διάρκεια του γεύματος στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών είχαμε μία εκτενή συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο αναφέραμε ότι πρέπει να έχουμε και κοινωνικούς δείκτες, να μην εξετάζουμε δηλαδή μόνο την, την ε, ανάπτυξη με ονομαστικούς όρους. Πρέπει να εξετάσουμε η ανάπτυξη αυτή, τι αντίκτυπο έχει στη ζωή των ανθρώπων. Πολύ χαίρομαι που η Πρόεδρος ε, ενδιαφέρεται να εργαστεί πάνω στο θέμα των δικτών. Η ανάπτυξη και η ευημερία δεν είναι αντίθετα, είναι θέματα που σχετίζονται μεταξύ τους. Ε, θέλουμε μία ολοκληρωμένη στρατηγική διαβίου μάθησης και η Φιλανδία θα το προωθήσει αυτό. Όσον αφορά τα δικαιώματα εργαζομένων, έχει υποβληθεί πρόταση για ελάχιστη αμοιβή αυτή βρίσκεται στο θεματολόγιο μας. Ε, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν επίσης έχει αναφέρει το θέμα αυτό. Προσβλέπουμε λοιπόν ε, με ενδιαφέρον ε, στις περαιτέρω εργασίες στο θέμα. Η κυρία Φοντερ Λάιεν αναφέρθηκε σε δύο τρόπους να προωθηθεί το θέμα, είτε συλλογικές συμβάσεις, είτε ε, κυβερνητικές ενέργειες. Όσον αφορά τις υποσχέσεις, η ανεργία των νέων είναι υπερβολικά υψηλή, χρειαζόμαστε δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στηρίξει δράσεις ε, στα κράτη-μέλη. Ε, έχουμε την εγγύηση για τους νέους, ένα θέμα στο οποίο ε, ήταν ιδιαίτερα δραστήρια η Φιλανδία. Ο προκάτοχός μου, ο κύριος Ιχαλάινεν, επένεσε την ε, εγγύηση για τους νέους και χαίρομαι που και η κυρία Φοντερ Λάιεν δίνει προσοχή στο θέμα αυτό και θεωρεί ότι πρέπει να αποτελεί τμήμα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Η Φιλανδία συμμερίζεται το στόχο αυτόν η εγγύηση για τους νέους και παρόμοιες δράσεις, μια γάμα από υπηρεσίες προς τους νέους θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τη Σουηδή συνάδελφο και άλλους που ανέφεραν το θέμα του ρατσισμού. Ο ρατσισμός απαγορεύεται σύμφωνα με την οδηγία κατά των διακρίσεων. Πρέπει να υπάρξουν δράσεις για την ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας. Τα συμπεράσματα θα επισημάνουν τα θέματα που σας ανέφερα. Χαίρομαι που είχα την ευκαιρία να απαντήσω έστω και σε λίγες από τις ερωτήσεις σας. Thank you. Κυρία Υπουργέ, είναι η σειρά σας να απαντήσετε τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις ερωτήσεις. Ήταν εξαιρετικές. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις περισσότερες από αυτές όσο το δυνατόν πιο γρήγορα δεδομένου ότι κατά την παρουσίασή μου Ήδη είπα σχεδόν τα πάντα. Θα προσπαθήσω και το ίδιο. Έκανα και το ίδιο και στις πρώτες μου απαντήσεις μετά από τον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Πάμε στο εξάμεινο. Σαφέστατα ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη τις προθέσεις της Κομισιόν επί του θέματος στο εξάμεινο. Θα πρέπει να εξελιχθεί ούτως ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το κοινωνικό πυλώνα. Επίσης αναφέραμε και άλλη μια φορά το πρόβλημα των αστέγων. Ήδη προηγουμένως ε, είπα, είπα ότι είναι αρμοδιότητα της Κρίστα Μίκονα, Υπουργού Περιβάλλοντος. Αλλά ε, σαφέστατα δεν είναι και ευχάριστο να ακούει κανείς ε, τέτοιες πληροφορίες ανησυχητικές Ελπίζω λοιπόν να καταφέρουμε να βρούμε μια λύση. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα μπορούσε να υπάρξει κάποια συμφωνία μεταξύ Κομισιόν και Γαλλίας επί του θέματος για να επιληθεί το πρόβλημα των αστέγων. Μετα, ε, αναφέρατε πολλοί από εσάς διάφορα προβλήματα ε, κενά τα οποία υπάρχουν. Πρέπει να γνωρίζετε ότι βρισκόμαστε σε μια στρατηγική φάση αυτή τη στιγμή. Και έτσι εξηγείται η ύπαρξη αυτών των ελλείψεων ε, συγκεκριμένων στοιχείων εδώ και εκεί. Το σημαντικό είναι στη συνέχεια να κάνουμε τα πράγματα πιο συγκεκριμένα, να αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την Κομισιόν. Σε στενή συνεργασία με την Κροατία και με τη Γερμανία τις επόμενες προεδρίες. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα σας ενημερώσουμε με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για να συνεχιστούν όλα τα θέματα που αναφέραμε σήμερα με στρατηγικό τρόπο. Ο άλλο στόχος, όπως ανέφερα, είναι η ευημερία, η, πρόθεση της ευημερία, της καλής διαβίωσης. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτως ώστε αυτό να γίνει πραγματικότητα στην Ευρώπη και με πολύ απτό τρόπο. Σαφέστατα δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Χρειαζόμαστε την υποστήριξη όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και τη δική σας υποστήριξη ούτω ώστε να διασφαλίζεται η ευημερία, η καλή διαβίωση στο σύνολο της Ευρώπης. Στην πρώτη μου ομιλία και όταν απάντησα στις πρώτες ερωτήσεις αναφέρθηκα στον Brexit και στον κανονισμό που υπάρχει επί του θέματος ε, από τις αρχές του χρόνου όπου διασφαλίζονται τα δικαιώματα και η κοινωνική προστασία των Βρετανών υπηκόων ακόμη και σε περίπτωση Brexit, όπως είπα προηγουμένως. Επίσης έχουμε μιλήσει για τη γύρανση, για τους ηλικιωμένου. Είναι σαφές ότι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι χρειάζονται φροντίδα, αλλά αυτό ενέχει ε, περιλαμβάνει και την αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εμείς δεν μπορούμε παρά να δράσουμε σε επίπεδο κρατών μελών. Το θέμα της ισότητας είναι ε, ιδιαίτερα σημαντικό. Ο Υπουργός Μπλουμφίντ ε, είναι αρμόδιος για το ζήτημα αυτό. Σαφέστατα σε επίπεδο Συμβουλίου θα γίνει πολιτική συζήτηση επί του θέματος, αλλά όχι πριν το Δεκέμβριο. Τώρα, ο, ο καρκίνος ε, στον επαγγελματικό χώρο. Αιτία θανάτων πολύ σημαντική ε, στην Ευρώπη περίπου 100.000 θανάτους προκαλεί η ασθένεια αυτή. Είναι ανατριχιαστικά τα νούμερα. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε τις προσπάθειες να ξαναδούμε τα διάφορα όρια που υπάρχουν, για παράδειγμα όσον αφορά τα διάφορα επαγγέλματα. Θα πρέπει λοιπόν να καθορίσουμε τις ε, οριακές τιμές ώστε να αποφευχθεί τόσο υψηλό ποσοστό θανάτων από επαγγελματικό καρκίνο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε τους προσκεκλημένους μας. Ε, θα ήθελα να τους ευχαριστήσω που παρευρέθηκαν στη συνεδρίασή μας και που απάντησαν όλες τις ερωτήσεις. Να ευχαριστήσω και τα μέλη για τις ερωτήσεις τους. Ε, αποτελούν απόδειξη τις ε, ειλικρίνες του ειλικρινούς τους ενδιαφέροντος ε, για συνεργασία με τη Φιλανδική Προεδρία. Εκ μέρους όλων μας θα ήθελα να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο για τη Φιλανδική Προεδρία και αναμένουμε με ανυπομονησία τη συνεργασία μας. Ευχαριστούμε. Ε, η Renew Europe έχει έναν βουλευτή παραπάνω από ό,τι χρειάζεται, ε, από ό,τι επιτρέπεται. Έχουμε τεχνικά προβλήματα, μήπως μπορεί κανείς να βοηθήσει, μήπως μπορείτε να, πάτε, να καθίσετε αλλού. Η Renew εξακολουθεί να έχει έναν παραπάνω βουλευτή. Όλα εντάξει τώρα, λήξη της ψηφοφορίας. result Το αποτέλεσμα είναι 43 ψήφοι υπέρ, 3 κατά, 3 αποχές. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγκρίθηκε λοιπόν το διορθωτικό. Το επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης ε, είναι τα διάφορα. Υπάρχει κανείς που να θέλει να πει κάτι. Κυρία Ζαλεύσκα, νομίζω ότι ξέρω τι θα πείτε. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Γραμματεία το επιβεβαίωσε ήθελα να πω ότι δεν ε, υπερεύει το χρόνο ομιλίας μου. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής μου, μου κλέψατε μισό λεπτό, Πρόεδρος. Είχαμε κάποια προβλήματα. και γι' αυτό δεν ε, ξαναξεκινήσαμε ε, το χρονόμετρο ε, όταν πήρατε το λόγο. Δεν φαινόταν ο πραγματικός ο χρόνος ομιλίας σας. Πράγματι, στο 1,5 λεπτό ήμασταν. σας παρακαλώ, δεχτείτε τη συγνώμη μου. Αυτά για σήμερα. Η ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης είναι... 3 ε, Σεπτεμβρίου, διότι έχει ακυρωθεί η 2η Σεπτεμβρίου. 3 Σεπτεμβρίου λοιπόν στις 9 το πρωί. Σας ευχαριστώ όλους σας και σας εύχομαι μια θερμή ημέρα. And the